για το Ιράν, για τη Σιρήνα και δίνω το λόγο στον κύριο Ματσάκη. Δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε που μόλις φτάσατε, η δίωξη της κυρίας Σιρήν Εμπάντη βραβείου Νόμπελ είναι μία από τις πολλές υποθέσεις που μας απασχολούν για το Ιράν αυτή τη στιγμή και αυτές οι διώξεις δεν αποτελούν έκπληξη για μας δεδομένου ε, του ότι υπάρχουν ε, αναχρονιστικές απόψεις ε, για τους κυβερνήτες αυτής της χώρας και δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι το καθεστώς στο Ιράν δεν θα λάβει καθόλου υπόψη του τα ψηφίσματά μας. Θα γελάσουν και θα τα πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο όπως έκαναν και για όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου μας. Και ποιος να τους κατηγορήσει. Γνωρίζουν ότι τα ψηφίσματά μας είναι μόνο λόγια και όχι πράξεις. Και στις, ε, κατά τις εκτιμήσεις τους ε, δεν αξίζουν τα καν το χαρτί πάνω στα οποία ε, τα τυπώνουμε. Για να φέρουμε κάποια αλλαγή στο Ιράν θα πρέπει τα λόγια μας να τα συνοδεύουμε δουλεύουμε με δράσεις, κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε το οποίο PMOI από τον κατάλογο των, τρομοκρατών μας, ή των τρομοκρατών μας ή να φροντίσουμε την σωστή συνεργασία ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών. Γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα μας πάρουν σοβαρά οι αρχές του Ιράν και θα το σκέφτονται περισσότερο ε, σε περίπτωση που θέλουν να ασκήσουν διώξεις κατά των πολιτών τους που υπεραμείνονται της δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε λοιπόν, κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε άλλο ένα ψήφισμα εκτός από αυτό εδώ που θα ζητά από τις κυβερνήσεις ορισμένων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως από την Βρετανία και από τη Γαλλία και από χώρες που θέλουν να γίνουν μέλη όπως η Τουρκία να σταματήσουν την υποκριτική τους στάση έναντι του Ιράν και να λάβουν άμεσα πραγματική δράση εναντίον του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. κυρία Στήλερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ιστορία της ε, Σίριν Αμπάντη, πρώτης γυναίκας ε, μουσουλμάνας που έλαβε το βραβείο Νόμπελ, που είναι και η πιο γνωστή για μας σήμερα. Ε, είναι η πρώτη γυναίκα δικαστή της χώρας της που αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω της Ιρανικής Επανάστασης. Υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών στο Ιράν, προσπαθώντας να αλλάξει την νομοθεσία σχετικά με το διαζύγιο και το κληρονομικό δίκαιο υπερασπίστηκε τις μειοψηφίες και τα δικαιώματά τους και πρόσφατα υπερασπίστηκε 7 μέλη του δόγματος Μπαχάη που είχαν συλληφθεί και που αντιμετωπίζουν διώξεις όπως και άλλα μέλη διαφορετικών ε, πεπιθήσεων στο Ιράν. Έχει το σεβασμό όλων μας ε, στο Κοινοβούλιο, διότι αυτοί μαζί με άλλους ε, Υπερμάχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ίδρυσαν το κέντρο υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο Ιράν και προσπάθησαν να υπερασπίσουν ε, τα θύματα ε, των διώξεων και τις οικογένειές τους. Οι αρχές προσπάθησαν να κλείσουν αυτό το κέντρο από την αρχή διότι θεωρούσαν ότι απειλούνταν. Τα μέλη του κέντρου υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δέχονταν απειλές και πολλές φορές εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια της κυρίας Ιρίνα Μπάντι. Και λίγο πριν από τα Χριστούγεννα λίγο μετά τα Χριστούγεννα, όταν ε, ήταν έτοιμοι να ε, εορτάσουν τη δέκατη επέτειο τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, έκλεισαν οι υπεύθυνοι του Ιράν το κέντρο υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητάμε λοιπόν από την Τσεχική Προεδρία και από όλα τα κράτη-μέλη να φροντίσουν να ανοίξει εκ νέου το κέντρο υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι δύσκολο για μας να καταλάβουμε την, το πραγματικό θάρρος που απαιτείται από υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η Σιρήνε Μπάντι για να μπορέσουν να δουλέψουν σε αυτές τις χώρες. Πρέπει λοιπόν να φωτίσουμε την κατάσταση που ισχύει στο Ιράν και να μπορέσουμε όλοι να δούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί γιατί αυτοί που προσπαθούν να βοηθήσουν ε, τους ε, αρρώσους και αναξιοπαθούντες κατηγορούνται ότι συνεργάζονται με ε, εχθρούς του καθεστώτος. Ο αγώνας ο δικός της είναι και δικός μας αγώνας και πρέπει να τη βοηθήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Λαμπέρ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Λάμπερτ. Είναι σημαντικό, πιστεύω, να βοηθήσουμε του υπερμάχου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε πιστεύουμε ότι θα μα ακούσουν οι κυβερνήσει, είτε όχι. Χρειάζεται μεγάλο ε, ε, θάρρο ε, για να ασκήσουν το έργο τους αυτοί οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα διότι πρόκειται για επιθέσει κατά μια υπερμάχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό δείχνει ότι δεν μπορούν να ασκήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους όπως ε, το δικαίωμα της, ε, των ελευθέρων πεπιθήσεων διαφορετικά διατρέχουν πολύ σοβαρό κίνδυνο. Η Σιρήνα Μπάντι ίδια πολλές φορές έχει αντιμετωπίσει απειλές ε, κατά της ζωής της διότι έχει υπερασπιστεί μέλη της, του δόγματος Μπεχάη στο Ιράν που υφίστανται σημαντικές διώξεις. Τις τελευταίες 24 ώρες ακολούθησαν και άλλες συλλήψεις ατόμων που συνεργάστηκαν με την κυρία κυρία και άλλων μελών του δόγματος Μπαχάη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι παρατηρούμε αυτή τη στιγμή μια αλλαγή στο πώ τα κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό έχει επιπτώσεις ε, και στις χώρες με τις οποίες έχει σχέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβόμαστε ότι δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι ε, φαίνεται ότι έχουμε εμπορικέ σχέσει με χώρε που δεν ε, δείχνουν να ενδιαφέρονται. Εμείς ε, θα πρέπει να δείξουμε ότι τηρούμε αυτές ε, ε, τις διατάξεις που έχουμε θεσπίσει και δεν θα πρέπει να ασκούμε, να έχουμε εμπορικέ σχέσεις με χώρες που δεν, τηρούν, δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε αυτούς που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκράτες που προσπαθούν να αμυνθούν κατά των μη δημοκρατικών καθεστώτων. Ευχαριστώ κύριε Κέλλον. δύο λεπτά ο συντάκτης και εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση των πολιτών ε, του Ιράν που ζουν υπό καταπιεστικές ε, συνθήκες του καθεστώτος των ε, μουλάδων είναι ανησυχητικές και συνεχίζουν να επιδεινώνονται από το 2005 σε όλους τους τομείς. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή να συνεχίσει την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και να υποβάλει μια πλήρη έκθεση της κατάστασης κατά το πρώτο εξάμεινο του έτους. Σήμερα διαμαρτυρόμαστε κατά των διώξεων κατά της κυρία Σιρίν Μπάντι, κατόχου του βραβείου Νόμπελ και υπερμάχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συχνά ε, ρωτάμε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το θέσουμε και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Το Ιρανικό καθεστώς ε, είναι δυνάμει μεγαλύτερη απειλή για το κράτος δικαίου και για την ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πολύ πιθανό ε, η κυβέρνηση του Ιράν να έχει ε, πυρηνικέ κεφαλέ και ήδη έχει πυράβλους με του οποίου μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να λάβουμε μέτρα γιατί ξέρουμε ότι το Ιράν υποστηρίζει τη Χεσμολά. δεν θα πρέπει να κάνουμε συμβιβασμού και δεν θα πρέπει να βοηθάμε ε, το καθεστώ τη, Τεχεράνης ε, να δένει τα χέρια τη αντιπολίτευση χαρακτηρίζοντα την τρομοκρατική οργάνωση. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή θέση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να θέσουμε ως προτεραιότητα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε φορά που συνελασσόμεθα με το Ιράν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μέγερ. Δύο λεπτά ο συντάκτης. Κύριε Πρόεδρε, η δίωξη της κυρίας Σέιν Μπάντι δεν είναι μεμονωμένη υπόθεση. Μεταξύ των υπερμάχων του καθεστώτος η κυρία Εμπάντι είχε μια προνομιούχο θέση και το Κέντρο Υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, διακηρύσει την ε, δραματική κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στο Ιράν. Διώκονται όχι μόνο άτομα για τις θρησκευτικέ τους πεπιθήσεις, αλλά και άτομα λόγω των σεξουαλικών τους πεπιθήσεων και πολλοί διακινδυνεύουν την φυλάκισή τους μπορεί να τους κοστίσει και τη ζωή τους ε, το ότι έχουν διαφορετικές ε, πεπιθήσεις. Ο εξωτερικός κόσμος ε, και η Ευρώπη δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται για αυτή την κατάσταση που είναι πραγματικά ανησυχητική, που θα έπρεπε να μας σοκάρει. Και οι διεθνείς κοινότητα ενδιαφέρεται για άλλα θέματα, ενδιαφέρεται για τη μείωση τη στρατιωτική δύναμη του Ιράν και για τη χρήση ατομική ενέργεια, ενώ θα έπρεπε να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα και να χρησιμοποιήσουμε ε, ε, ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας ε, και τι εμπορικέ μα σχέσει, για να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να δεχθούμε αυτό το έλλειμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι πιο σημαντικές ομάδες της αντιπολίτευσης είναι στο κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων πολλών χωρών της Δύσης και αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Η κυρία Μπάντι είναι ένα από τα θύματα του καθεστώτος του Ιράν είναι ε, ιδιαίτερα γνωστή και το ότι είναι κάτοχος του βραβείου Νομπέλ της είχε διασφαλίσει την ε, ε, ελευθερία της μέχρι τώρα. Θα πρέπει να λάβουμε κατεβηγόντως μέτρα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόσελτ, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το γραφείο μου στο Μόναχο βρίσκεται σε ένα δρόμο στον οποίο βρίσκονται πολλοί χριστιανοί Αρμένοι από το Ιράν ανήκουν ε, σε μία από τις παλαιότερες χριστιανικές κοινότητες ε, του κόσμου και είναι και ε, πατριώτες της χώρας τους, του Ιράν ενοχλούνται από την μυθαλλοδοξία έναντι των πολλών θρησκευτικών κοινοτήτων και δεν είναι ίδιον της χώρας τους. Θεωρούν ότι είναι αντίθετο με τις παραδόσεις ενός από τα παλαιότερα κράτη της γης. Δεν είναι αντίστοιχη με τις παραδόσεις τους η στάση των μουλάδων. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Η κυρία Σινεμπάντι από τότε που έλαβε το, γραφείο, το βραβείο Νόμπελ ε, διατρέχει πολύ σημαντικού κινδύνους, ε, κινδύνου που διατρέχουν και τα μέλη όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων διώκεται και χρειάζεται επιγόντως την αλληλεγγύη μας. Κάνω έκκληση λοιπόν προς την ε, Προεδρία του Συμβουλίου που ασκείται από την Τσεχία να στραφεί άμεσα προς την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Ευχαριστώ. Κύριο Σπίνιορ, δύο λεπτά εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταρχάς θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της τσεχικής προεδρίας παρόν. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι κρίμα, ε, είναι αμαρτία που δεν υπάρχει κάποιος εδώ εξ της τσεχικής ε, ε, προεδρίας, γιατί υποτίθεται η προεδρία είναι ένας από τους βασικούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. κατά διάρκεια της γερμανικής προεδρίας δεν είχαμε τέτοιου είδους προβλήματα. Το Ιράν είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Μία από τις χώρες που έχει έναν βαρύνοντα λόγο για το μέλλον της ε, περιοχής. Γι' αυτό θα πρέπει και οι Ιρανικές αρχές να σεβαστούν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, τους ανθρωπιστικούς ε, νόμους. Εδώ είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα της κυρίας Σιρίν Εμπάντη, η οποία έχει κερδίσει και το, της έχει απονεμηθεί και το βραβείο Νόμπελ. Η δίωξή της προφανώς ε, είναι αστήρικτη εδώ έχουν ε, συλληφθεί φοιτητές του Πανεπιστημίου Σιράζ και άλλοι έξι φοιτητές ε, στις 12 Ιανουαρίου συνελήφθησαν. Επομένως θα πρέπει να δώσουμε μία μάχη όχι μόνο για την κυρία Μπάντι αλλά και για τους φοιτητές ε, της Περσίας, του Ιράν. Επίσης διώκονται και γιατροί οι οποίοι κάνουν τεστ για το AIDS. Πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούτοβιτς έχει ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Το Ιράν είναι μια χώρα φονταμενταλιστών κατά βάση, αλλά και δημοκρατικών θεσμών μάλλον και να μιλήσουμε για δημοκρατικούς θεσμούς είναι κάτι το οποίο δεν έχει, δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Η πολιτικοί του Ιράν θέλουν να φαίνονται ότι είναι προοδευτικοί, θέλουν να φαίνονται ότι είναι δημοκρατικοί, εξού και προσυπογράφουν διάφορες διεθνείς συμβάσεις, αλλά επί της ουσίας πω όσοι ενδιαφέρονται για τις, για τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Και βλέπουμε εδώ την ε, δίωξη της κυρίας Σιρίν Εμπάντη. Εμείς υποστηρίζουμε πλήρως το ψήφισμα, έστω και αν θεωρούμε θα έπρεπε να είναι πιο ριζοσπαστικό. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία του Catch the Έχουμε τρεις ε, υποψηφίους. Ο κύριος Ναζαρέ. Ε, εάν είστε γρήγοροι θα μιλήσετε και οι τρεις, αλλιώς οι δύο. Αυτή είναι μία από τις ε, λιγότερο γνωστές ε, ε, περιπτώσεις δίωξης και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκτός όμως από την περίπτωση της κυρίας Εμπάντη έχουμε και τους φοιτητές οι οποίοι διώκονται και συλλαμβάνονται. Ε, χαίρομαι που το ψήφισμα αυτό έχει προσυπογραφεί από διάφορες, από όλες τις ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προέρχομαι από μια χώρα που ήταν στο παρελθόν κομμουνιστική και δεν ε, ήταν διασφαλισμένη η ελευθερία της έκφρασης στη χώρα μου. Γι' αυτό ελπίζω ότι θα μπορέσουμε ίσως κάτι να κάνουμε στην περίπτωση του Ιράν. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω πλήρω το ψήφισμα, αλλά πιο συγκεκριμένα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τους συναδέλφους όπως ο κύριος Ματσάκης που είπαν ότι το βασικό πρόβλημα είναι η πολιτική καθησυχασμού αν θέλετε που έχουμε απέναντι στην κυβέρνηση της, ε, του, του Ιράν. Δηλαδή ο σεβασμός δικαιωμάτων, δικαιωμάτων ε, μπαίνει σε μια δεύτερη με, μοίρα. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, πραγματικό πρόβλημα και εμείς ε, το κρύβουμε αυτό για να προωθήσουμε μία πολιτική ε, που ευνοεί ε, την δημιουργία τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Μουτσαχεντίν που από τη μια πλευρά τους βάζουμε σαν, σαν τρομοκρατική οργάνωση και από την άλλη συνδιαλεγόμεθα μαζί τους. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μπρεζίνσκι πιστεύει ότι μία από τις ε, μεγαλύτερες ε, απειλές ε, που αντιμετωπίζουμε είναι οι σχέσεις των χωρών στη Μέση Ανατολή και κυρίως και πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να επιληθούν τα προβλήματα στην περιοχή εάν τυχόν δεν εκδημοκρατιστεί το Ιράν. Όμως ο εκδημοκρατισμός δεν πρέπει να γίνει εκ των ε, έξω, εκ ε, έξω αν θέλετε, εκ των έσω πρέπει να γίνει αυτό. Και προφανώς βέβαια χρειάζεται και ο κόσμος την υποστήριξή μας. Γι' αυτό θα πρέπει να, να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε δημοκρατική ε, δύναμη σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Α, και ένας τέταρτος συνάδελφος ζήτησε το λόγο. Ο κ. Ζαλεύσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ηρωνικά θα έλεγα ότι όπως και στην Χαμάς η, και εδώ οι, οι, αρχές ε, είναι αποτέλεσμα εκλογών, ε, λαϊκής θέλησης και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα διότι μπορούμε να πούμε τις απόψεις μας, ε, μπορούμε να πούμε ότι καταδικάζουμε την πολιτική τους συναφορά, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω και τα λόγια μας ίσως γίνουν τα όπλα μας και να υποστηρίξουμε αυτούς που συνεχίζουν να υπερασπίζονται την ελευθερία στο Ιράν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, δεν ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό. Ο κύριος Σπίτλα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης της κυρίας Σιρήν Μπάντι και θεωρεί ότι οι απειλές ε, τις οποίες δέχεται και η ίδια και η συναδελφή της, ιδιαίτερα μετά την έρευνα που έγινε στο γραφείο της στην Τεχεράνη στις 29 Δεκεμβρίου, είναι απολύτως απαράδεκτες. Η έρευνα στο γραφείο της ε, είναι ε, η τελευταία πράξη εκφοβισμού που έχει γίνει κατά της κυρίας Σινεμπάντη και σε αυτές τις πράξεις εκφοβισμού συμπεριλαμβάνονται, συμπεριλαμβάνεται η αναστολή των δραστηριοτήτων ε, του Κέντρου Υπεράσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, του οποίου προήσατε η κυρία Εμπάντη. Υπάρχουν δύο ψηφίσματα, δύο δηλώσεις της 31ης ε, Δεκεμβρίου πέρυσι της 21ης συγγνώμη, Δεκεμβρίου πέρσι και ε, η Επιτροπή πιστεύει ότι θα πρέπει να τηρούνται να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα του συνέρχεστε, το οποίο περιλαμβάνεται στη Διεθνή Πράξη Πολιτικών Δικαιωμάτων που έχει υπογράψει και επικυρώσει το Ιράν. Και θα πρέπει η κυβέρνηση του Ιράν να ε, επανεπιτρέψει το άνοιγμα του Κέντρου Υπεράσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να χορηγήσει το νομικό καθεστώς το οποίο ζητείται για το κέντρο αυτό τα τελευταία χρόνια. Το 2009 η Επιτροπή θα προσπαθήσει σε κάθε ευκαιρία ε, να ασκήσει πίεση έναντι των αρχών του Ιράν, ούτως ώστε να δοθεί στην κυρία Εμπάντη και σε άλλους επεμβάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο Ιράν η ελευθερία να δράσουν στη χώρα χωρίς εκφοβισμούς και απειλές. Όπως ε, γνωρίζουμε όλοι, τα θέματα της ε, πυρηνικής ενέργειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιορίζουν το πεδίο των σχέσεών μας με το Ιράν. Θα συνεχίσει η Επιτροπή να δράσει στον τομέα κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Έχουμε επίσης κατορθώσει να διατηρήσουμε κάποια προγράμματα που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την χρηστή διακυβέρνηση, όπως επίσης και την ε, το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών, κάτι που κάνουμε μαζί με τη UNICEF ε, και το θέμα της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος. Ακόμη προσπαθούμε ε, να βελτιώσουμε ε, τομείς όπως η παιδεία και ο πολιτισμός. Στο πλαίσιο του Εράσμους Μούντους είχαμε μια επίσκεψη Ιρανών δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες και υποστηρίζουμε και την εκπομπή προγραμμάτων και εκπομπών στην περσική γλώσσα. Παρ' όλα αυτά είναι σαφές ότι αν ε, δεν αλλάξει η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, δεν θα μπορούν να εξελιχθούν φυσιολογικά οι σχέσεις μας με τη χώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μόλις τελειώσει η συζήτηση θα γίνει η ψήφιση αυτής της εκθέσεως. Και τώρα έχουμε ε, το ψήσμα για την Γουινέα Συμφωνία Διάταξη. Ο κ. Ματσάκης έχει το λόγο για δύο λεπτά. Mr. President, Mr. Commissioner. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ιουνέα έχει γνωρίσει μια πολύ ιστορία, διότι έχουμε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες συνεχώς